Colleagues, please take... Ναι, συνάδελφοι, καθίστε. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση. Ξεκινώντας θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών φυσικά και την ΣΕΜΑ της Λετωνίας, την το Κοινοβούλιο της Λετωνίας που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων όπως λέμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη συνάντησή μας. Η συνάντησή μας αυτή είναι τμήμα της διαδικασίας ε, της Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας όπως τη λέμε και νομίζω ότι είναι και ένα από τα βασικά στοιχεία, από τα βασικά τμήματα αυτής της διαδικασίας που μας επιτρέπει να έχουμε έναν άμεσο διάλογο για συγκεκριμένα θέματα. Θέματα τα οποία πράγματι απαιτούν στενή συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε εντοπίσει δύο κυρίως θέματα και γι' αυτό έχουμε δύο τμήματα στη συνεδρίαση όπως ξέρετε. Το πρώτο αφορά στις νέες μορφές ε, συντονισμού εναντίον της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και το δεύτερο είναι δημοκρατικός έλεγχος των εποπτικών αρχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να σας πω ότι μιας και είμαστε πάρα πολλοί οι συμμετέχοντες σε αυτήν την συνεδρίαση, δεν θα είναι δυνατόν να πάρει το λόγο όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε ε, πάρα πολλά κοινοβούλια. Δύο λεπτά θα μιλήσει ο εκπρόσωπος του κάθε κοινοβουλίου εφόσον το επιθυμεί και θα δούμε πώς ε, θα προχωρήσει η συνεδρίαση. Έχετε κάρτες μπροστά σας για να ζητάτε το λόγο. Γενικότερα θα προχωρήσουμε σύμφωνα με την εξή διαδικασία. Τρεις εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων, ένας Ευρωβουλευτής, αυτή θα είναι η διαδικασία. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο εντοπίσαμε τα συγκεκριμένα αυτά θέματα σαν έχοντα μεγάλη σημασία. Ξέρετε ότι θα ξεκινήσει και μια διαδικασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, θα δούμε ποια θα είναι η μορφή της, αλλά εμείς σαν ΕΚΟΝ, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, θα ξεκινήσουμε με μια έκθεση πρωτοβουλίας νομοθετική, και θα προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε τα προβλήματα και τους τομείς στους οποίους μια πλήρης νομοθετική πρόταση μπορεί να προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσουμε τη νομική πλαισίωση της φορολογίας γενικότερα. Σχετικά τώρα με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τον ρόλο ε, των κρατών μελών, θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να συζητήσω μαζί σας, να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Θα δώσω το λόγο τώρα για τρεις σύντομες εισαγωγικές ομιλίες, πέντα λεπτού η καθεμία. Ο κύριος Μπάλτς έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω για αυτή την πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα των εταιρικών φόρων είναι σημαντικό. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι θέμα που μας απασχόλησε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική εντολή και η συζήτηση θα εντατικοποιηθεί και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο η σκιώδης οικονομία στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, καλύπτει περίπου το 1 πέμπτο του ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού. Σε ετήσια βάση το κόστος αυτών των απαράδεκτων πρακτικών φτάνει το 1-3 ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα αυτό είναι αντιδιοντολογικό και άδικο για αυτούς οι οποίοι εργάζονται σκληρά και συνεισφέρουν με δίκαιο τρόπο στους φόρους και επιτρέπουν στην κοινωνία να λειτουργήσει σωστά και είναι κάτι που στερεί τεράστια ποσά από το μίσο όπως η ε, κοινωνική κάλυψη, τα σχολεία, η υγεία κτλ. και δημιουργεί στρεβλά περιβάλλοντα λειτουργίας των επιχειρήσεων και θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες των χωρών μας να αποκαταστήσουν τα δημοσιονομικά τους η φοροδιαφυγή και η φοροαποφύγη υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη και στη δημόσια διοίκηση. Έχει σημασία να υπογραμμίσουμε εδώ ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις απάτες τις φορολογικές και στη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή είναι κάτι ε, το οποίο ε, μπορεί να γίνεται και σε εισαγωγικά νόμιμα μέσω της παράνομης χρήσης των νόμιμων διαδικασιών. Ενώ ε, η απάτη φυσικά είναι η απλά μη πληρωμή των φόρων. Υπάρχει λοιπόν εδώ χώρος για ενίσχυση της συλλογικής μας ικανότητας να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Όλες οι χώρες θίγονται από το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και θέματα διαμεθοριακά επίσης που απαιτούν διαμεθοριακές λύσεις για να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε μια αποτελεσματική μορφή καταπολέμησης ε, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Θέλουμε οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εντάξει με τις φορολογικές τις υποχρεώσεις σε όλες τις χώρες μέλη στις οποίες δραστηριοποιούνται. Αυτό θα αυξήσει θα βελτιώσει τα δημοσιονομικά των χωρών μελών και θα επιτρέψει οι πολίτες να έχουν καλύτερες δημόσιες παροχές και υπηρεσίες. Το θέμα θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπιστεί με σωστό τρόπο. Η καταπολέμηση αυτών των φαινομένων θα περνισμένο τρόπο και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα σήμερα όπου οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ε, διασυνδεδεμένες και ταυτόχρονα πάρα πολύ διαδεδομένες και ευκίνητες. Υπάρχει ο φορολογικός ανταγωνισμός που δίνει κάποιες δυνατότητες εξυγχρονισμού και βελτίωσης των φορολογικών συστημάτων. Σύμφωνα με το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες εδώ περιορίζονται στις διαδικασίες χαμηλού επίπεδου κάτι το οποίο δίνει ε, υψηλά επίπεδα επικουρικότητα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες των ε, κρατών μελών έτσι ώστε να ε, γίνουν οι φορολογικές τους διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, πιο δίκαιες, αφαιρώντας απαράδεκτες εξαιρέσεις, αδικίες και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συλλογής των φόρων έτσι ώστε να ενισχυθεί η πολιτική καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα και της μεταφοράς κερδών σε τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιστεύει ότι θα πρέπει να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις οι οποίες να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της επιχειρηματικής κανότητας και του καθορισμού των φορολογικών ρυθμίσεων. Η Επιτροπή μας θα συντάξει την έκθεση αυτή και όπως είπα στην αρχή θα έχει σαν στόχο την βελτίωση κυρίως της διαφάνειας και της σύγκλησης στον τομέα ε, του φόρου επιχειρήσεων. Ε, ταυτόχρονα έχουμε ε, εδώ αναμένουμε πολλά και από την ομάδα των 20 Ε, η οδηγία η οποία αυτή τη φάση βελτιώνεται ε, προβλέπεται να κατατεθεί η πρόταση σε λίγο καιρό και η Ένωση θα γίνει ηγέτης, ε, θα έλεγα, σε επίπεδο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογουμένων. Ε, η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο τον προηγούμενο χρόνο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ήταν κάτι το πάρα πολύ θετικό και στην ε, ομάδα του Συμβουλίου αλλά και στην ομάδα ε, της, των 20. Αυτή η ανταλλαγή θα πρέπει να γίνει σε αμοιβαίο επίπεδο και να μην περιοριστεί στην ομάδα των 20, στο G20, Και εδώ τίθενται βέβαια και το θέμα ε, της ε, επικουρικότητας, ε, το οποίο επιτρέπει στις χώρες να παίρνουν επιμέρους μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι οδηγίες οι ισχύουσες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με στρεβλό τρόπο με στόχο την αποφυγή πληρωμής φόρων και θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας λοιπόν προς τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή έτσι ώστε να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο ε, μέσο ε, ε, αποτροπής τέτοιου είδους απαράδεκτων φορολογικών συμπεριφορών. Το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια σωστή βάση για μια έλογη συνένεση στην παρούσα φάση το Κοινοβούλιο δημιουργεί μια επιτροπή έρευνας σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές στον τομέα της φορολογίας. The extension of the automatic exchange of information on tax rulings. Να υπάρξει σωστή ενημέρωση για τις αποφάσεις αυτές από τις διάφορες χώρες και νομίζω ότι ήδη από την Άνοιξη θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Νομίζω ότι η προσπάθεια καταπολέμησης αυτών των απαράδεκτων φαινομένων θα πρέπει να είναι βασικός στόχος μας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Και γι' αυτό και η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι κάτι το θετικό. Έχουν πολλά να πούν τα εθνικά κοινοβούλια και αυτό ακριβώς υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινή πρόοδο και για καλύτερο συντονισμό στον τομέα της φορολογίας. Thank you very much. I give the floor. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούρκαρτ, επόμενος ομιλητής η Ανελής Ντότς. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πεπειραμένους βουλευτές και πολυάριθμους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συνάντηση και περιμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Πέντε λεπτά ε, είναι ο χρόνος αγόρευσης ε, ημών εδώ στο πάνελ για να έχουμε πραγματικά χρόνο για συζήτηση. Και αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι είναι σαφές για όλους τους βουλευτές ότι η πρόληψη να υπάρχει ένας κίνδυνος ε, με τον εκθετικό φορολογικό σχεδιασμό, τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, είναι προς το δικό μας συμφέρον. Διότι αν αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, θα δούμε μεγάλη αγανάκτηση, όπως είδαμε ήδη μετά την υπόθεση με το Λουξεμβούργο και τις τράπεζες διαδικασίας LAX, το ίδιο θα, θα δούμε και μάλιστα ε, θα δούμε να αυξάνεται αυτή η αγανάκτηση. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν σε για παράδειγμα, οι, οι απλοί άνθρωποι που λένε ότι πρέπει να πληρώσουν το φόρο ε, και πρέπει να τηρήσουν στο έπακρο τι ε, δεσμεύσει τους και κάποιοι άλλοι μπορούν να φοροδιαφεύγουν, να φοροαποφεύγουν. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε ε, την αξία της πολιτικής και των πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε πολύ ότι είναι η Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας. Όλοι όμως οι πολιτικοί νομίζω ότι έχουμε αυτή την τελευταία ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε ε, τις αθέμητες φορολογικές πολιτικές σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Πρέπει ε, τις ε, πολιτικές να τις ξεπεράσουμε. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που δεχτήκατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα από κοινού γιατί δεν νομίζω ότι είναι κομματικό θέμα. Και ο κύριος ε, Μπούλτ, συνάδελφος, είπε πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Και πράγματι πολλά κόμματα συμφωνούν, επί της αρχής τουλάχιστον. Και το έχουμε δει σε πολλές διαφορετικές ε, πτυχές ε, που αφορούν την εταιρική φορολογία. Ένα παράδειγμα το είπε και ο κύριος Μπουλτ. Είναι αυτή η κοινή ενωπημένη φορολογική βάση. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι πρέπει να είναι πιο ξεκάθαροι οι ορισμοί των φορολογητέων στοιχείων, ε, περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων. Και σε επίπεδο ΣΑ έχουμε κάποιους κανόνες, όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και όποτε ερχόμαστε πιο κοντά στο θέμα της εφαρμογής αυτών των ε, κανόνων και ζητημάτων, βλέπουμε ότι κάποιες φορές ο σημασίας ε, διαφορές ερμηνείας τελικά συγκρατούν κάποιες κινήσεις θα πρέπει εμείς οι βουλευτές να δείξουμε ότι η δημοκρατική πολιτική προσέγγιση ε, είναι μια καλή πολιτική για να υπερπηδήσουμε τις διαφορές τις εθνικές. Δεν μπορεί να είναι σωστό οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληρώνουν τους φόρους τους και να υπάρχουν κάποιες εταιρείε εντός Ευρώπης οι οποίες να μπορούν να πληρώνουν γύρω στο 1 ή και λιγότερο της 100 εταιρικό φόρο. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό ως βουλευτές, επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να λάβουμε μέτρα. Ε, είναι πολλά από αυτά εδώ και καιρό επιτάπητος, ε, σχεδιάζονται και πολλοί βουλευτές ε, στα κοινοβούλια σας έχετε ζητήσει να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την κοινή, την ενιαία φορολογική βάση. Επίσης πρέπει να έχουμε ένα κοινό ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Να το λύσουμε επιτέλους αυτό το ζήτημα. Πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό, δεν ξέρω, ένα μαύρο κατάλογο εταιριών ίσως για όσες εταιρείε ε, έχουν ε, πραγματικά ε, προβεί σε φορολογική αποφυγή και να δούμε και ποιοι σύμβουλοι τους βοήθησαν. Υπάρχουν και μέτρα για την υποβολή εκθέσεων των κερδών από τις πολυεθνικές. Για το τραπεζικό τομέα ισχύει αυτό και είναι καλό. Πρέπει να το δούμε για τις πολυεθνικές όμως επίσης. Και τι μέτρα, τι μηχανισμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα και μάλιστα γρήγορα. Γιατί οι ψηφοφόροι αυτό ζητούν από εμά και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αυτό ζητούν από εμά. Ω βουλευτέ, επίση, θα πρέπει να φροντίσουμε οι συζητήσει, ο διάλογο, η διαδικασία, η πολιτική για τη φορολογία να ε, συμπεριλάβει όσο δυνατόν περισσότερε πλευρέ. Λέγεται ότι η φορολογική πολιτική δεν περιλαμβάνει ε, του κοινωνικού εταίρου στο βαθμό που θα έπρεπε. Ότι δεν αντιπροσωπεύονται όλοι οι κλάδοι οικονομική δραστηριότητα, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνδικαλιστέ, κοινωνικών πολιτών. Και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Είμαι βέβαιη ότι περισσότεροι στην αίθουσα θα συμφωνούσαν. Πρέπει να υπερβούμε απλά και μόνο τη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Κάτι παραπάνω θα μπορούσε να είναι επώδυνος μέτρο. Όμως όλοι όσοι συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα και ιδίω ε, που είναι στην κυβέρνηση, θα πρέπει να δεχθούμε την υπευθυνότητα, την ευθύνη που έχουμε. Μπορεί να μην είμαστε πάντα ε, προβλεπτική. Δεν δρούσαμε πάντα ε, προκαταλαμβάνοντας κάποια πράγματα. Όμως αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που ζητούν οι πολίτε και πρέπει να του παρέχουμε και το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τι μικρομεσαίε επιχείρησει, το οποίο ο κύριο Μπούλτ. Και αυτό πρέπει να το πετύχουμε. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Οι πιο επιτυχημένε εταιρείε θα είναι αυτέ που προσφέρουν ε, τα πιο ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίε. Και όχι αυτέ που θα έχουν του πιο ευφυεί ε, φορολογικού συμβούλου. Προσβλέπω λοιπόν να, να έχουμε μια καλή συνεργασία με όλες και όλους εσάς στο μέλλον, να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και ένα διάλογο καλό και τους επόμενους μήνες. Λίγους μήνες όμως, όχι πολλούς, γιατί πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Thank you. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανελίζ. Ο κύριος Βαλέρ Μουταριέ είναι ο επόμενος, θα λάβω το λόγο, είναι η διευθυντή στην ΚΑΜΑ Τάξουντ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ αυτό το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ σήμερα να πάρω το λόγο εδώ. Ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας πω δύο λόγια για το ποια είναι η δική μας δέσμευση σε αυτήν την προσπάθεια. Και εγώ συμφωνώ απολύτως ότι πραγματικά πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα, το θέμα είναι πολύ επίκαιρο. Ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ και ο επίτρος Μοσκοβίση έχουν θέσει το θέμα αυτό στην καρδιά των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και ήδη έχουμε ξεκινήσει σοβαρές προσπάθειες για την καταπολέμηση της ε, φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής ήδη από το 2012, το πρόγραμμα του 2012, κάτι που έχει οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Βεβαίως, εάν γίνει διάκριση μεταξύ του φορολογικού σχεδιασμού, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φορολογικής απάτης, πολλά θα πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχει επεξεργαστεί όσα και το G20. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες φορολογικές πρακτικές, οι οποίες ναι μεν είναι νόμιμες, δεν θεωρούνται όμως πλέον ε, πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει λοιπόν το 2015, και αυτό είναι μάλιστα και γεγραμμένο στο πρόγραμμα εργασιών μας, μία προσπάθεια όσον αφορά την διαφάνεια, την φορολογική διαφάνεια και δεύτερον όσον αφορά τον ε, ίσο φορολογικό ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική συνεργασία, η ενισχυμένη διοικητική συνεργασία με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, όπως είπε και ο κύριος Βάλς, είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πολύ σημαντικά προχωρήσει με την άρση του τραπεζικού απορρίτου, με την αυτοποιημένη ανταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών και φορολογικών πληροφοριών. Έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες, το Άγιο Μαρίνο, την Ανδόρα, το Μονακό, το να και την Ελβετία. Όσον αφορά τη διαφάνεια, βεβαίως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε ξεκινήσει με τις περίφημες tax rulings, τις φορολογικές αποφάσεις, αλλά βεβαίως όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή φορολογικών αποφάσεων, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει και τα κράτη-μέλη περιμένουν πολλά από μας, καθότι θεωρούμε ότι πολλά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι μια καλύτερη συνεργασία θα οδηγήσει σε πολύ πιο ορθή και δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων ε, στις χώρες που βρίσκονται. Όσον αφορά το φορολογικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, η προσέγγιση μας για το θέμα αυτό είναι περισσότερη συνεργασία έτσι ώστε η φορολόγηση των επιχειρήσεων να λαμβάνει χώρα εκεί όπου λαμβάνει χώρα η πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Καθότι σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν μεταφορά, μεταφορές κερδών εκεί όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι πιο ε, συμφέροντες για τις επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θέλουμε να καταργήσουμε εντελώς τον φορολογικό ανταγωνισμό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υπάρξει συσχετισμός μεταξύ της φορολόγησης και του τόπου στον οποίο λαμβάνει η χώρα η οικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Βεβαίως έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες που έχουν αποφέρει αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η σχέση μεταξύ της έδρας και των θηγατρικών, η αποφυγή της διπλής φορολόγησης και η Προεδρία της Λετωνίας έχει δεσμευθεί σε αυτούς τους τομείς ιδιαίτερα όσον αφορά την οδηγία για τους δασμούς και τα τέλη και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας έτσι ώστε να δούμε πώς οι συμφωνίες που υπάρχουν θα μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο με διαφάνεια για να διασφαλίσουμε την νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις μας και για τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει στο πρόγραμμα εργασιών της μία πρωτοβουλία για το επόμενο εξάμεινο έτσι ώστε να επανεξετάσει την φορολογία των επιχειρήσεων καθώς και την εγγύηση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Θέλουμε επίσης να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει μια νέα, πιο δυναμική συζήτηση, διαπραγμάτευση όσον αφορά τα θέματα αυτά της ε, φορολόγησης των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μας τη δυνατότητα να μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε όλη την εσωτερική αγορά, να μειώσουν το διοικητικό, το φορολογικό άχθος, να ξεπεράσουν σημαντικές δυσκολίες έτσι ώστε το σύστημα να γίνει λιγότερο περίπλοκο και πιο δίκαιο. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι οι βασικοί φορείς για τις αποφάσεις σε θέματα φορολογίας συνεχίζουν να είναι τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια, καθότι η αρμοδιότητα σε μεγάλο βαθμό παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Γι' αυτό και η κάθε κοινοτική δράση βεβαίως θα πρέπει να συμπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να οδηγηθούμε σε φορολογικά συστήματα τα οποία θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Δεν θα επανέλθω εδώ στις βασικές αρχές της ανάλυσής μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η φορολόγηση της εργασίας να είναι τόσο ε, βαριά και θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις που θα κατευθύνουν τη φορολογία έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η ανάπτυξη, ένα σύστημα λιγότερο περίπλοκο, να οδηγήσουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες πιο ευνοϊκό για την απασχόληση και για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το πνεύμα στο οποίο εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασιζόμαστε τα Εθνικά Κοινοβούλια στην στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως ε, βλέπουμε πόσο ενδιαφέρουσες είναι οι συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο παρόλο που πολλές φορές θεωρούμε τον ρυθμό υιοθέτηση αυτών των αποφάσεων λίγο απογοητευτικό. Αυτό βεβαίως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι χρειάζεται ομοφωνία για να ληφθούν αποφάσεις ε, για θέματα φορολογίας. Θα Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω αυτά που έχετε να πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρώτος ομιλητής είναι από το Κοινοβούλιο της Λετωνίας, ο κύριος Μέλτενς. Έχουμε 12 ομιλητές. Ο καθένας ε, θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μείνω στα δύο λεπτά. Η συστηματική αντιμετώπιση των φορολογικών απατών είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Η Λετωνία και στα πλαίσια της Προεδρίας ακολουθεί το λεγόμενο BPS και τα θέματα BPS. Προτεραιότητα της Λετωνικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι η περαιτέρω επεξεργασία φορολογικών ρυθμίσεων, νομοθετικών συγγνώμη ρυθμίσεων που θα έχουν σαν στόχο την ε, μείωση του φαινομένου των φορολογικών απατών και της φοροδιαφυγής. Τίθεται και το θέμα των ειδικών tax rulings ε, περιπτώσεων. Η Προεδρία της Λετωνίας θα υποστηρίξει την προσπάθεια την οποία, ε, η οποία ξεκίνησε μέσω της του κώδικα συμπεριφοράς έτσι ώστε να είναι σεβαστά και συμβατά τα περιεχόμενα των νομοθετικών ρυθμίσεων. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πλήρως την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία η οποία τροπολογήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, είναι ένας από τους στόχους της Προεδρίας μας. και αυτό αφορά και στην οδηγία για την αποταμίευση. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των επιμέρους περιπτώσεων εισοδημάτων. Οι προκλήσεις όμως παραμένουν να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες οι οποίες βρίσκονται υπό εξέταση στην παρούσα φάση και οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες και μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση. Θέματα όπως το ελάχιστο ποσοστό φορολογίας. Είναι κάτι το οποίο είναι θέμα αρμοδιότητας εθνικής. Τώρα η πρόταση συγκεκριμένη για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Λετωνία θέλει να συνεχιστεί η προσπάθεια η οποία γίνεται σε σχέση ε, με την κοινή ενοποιημένη βάση και να εξεταστεί η συμβατότητά της με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Λετωνία, όπως και άλλες πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν θέματα επίσης και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροδιαφυγής σε εθνικό επίπεδο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει με την πρωτοβουλία μηδενικής δήλωσης, όπως επίσης και με ένα πρόγραμμα εκ των υστέρων που ονομάζεται Αμνηστία Φορολογική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας κάποιος φορολογικός ανταγωνισμός και απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπερζέ από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις που θα αφορούν και δεν θα σας εκπλήξει αυτό ε, τα tax rulings, αυτές τις φορολογικές συμφωνίες. 26 συμφωνί, ε, μάλλον ε, χώρες εφαρμόζονται αυτού του είδους συμφωνιών εδώ και χρόνια, 20 τουλάχιστον νομίζω, με διάφορα μοντέλα, διαφορετικά από μια χώρα στην άλλη, μπορώ να σας ε, δώσω ε, πολλά παραδείγματα γιατί δεν έχω χρόνο. Το βασικό όμως ότι λαμβάνονται εκ των ε, πρωτέων κάποιες αποφάσεις, μονομερείς αποφάσεις είναι, μιας εθνικής φορολογικής διοίκησης. Δεν πρόκειται για μια σύμβαση ούτε για μια συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η πρακτική των tax rulings. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτή η πρακτική με απάτη. Για λόγους που μου διαφεύγουν, έχει ε, μπει στο στόχαστρο ε, αυτών των αποφάσεων τις τελευταίες εβδομάδες στο Λουξεμβούργο με την υπόθεση LuxLeaks και τα λοιπά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Μεγάλο Δουκάτο κάνει ακριβώς αυτό που κάνουν και τα άλλα 25 κράτη με αυτές τις νόμιμες ε, πρακτικές φορολογικών συμφωνιών τύπου tax ruling. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Άρα πρόκειται για μια πρακτική σύμφωνη με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και σύμφωνο με τους κανόνες περιδιπλής φορολογικής. Ίσως ενδεχομένως μεταξύ, η σχέση μεταξύ κανόνων και πρακτικών, ε, μεταξύ των διεθνών κανόνων ή ε, συμβάσεων περί μη φορολόγησης μπορεί να οδηγήσουν σε αποφάσεις με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και αυτό να θεωρείται ε, από ηθικής πλευράς ίσως όχι τόσο αποδεκτό. Αν συμφωνούμε από αυτού, ας αλλάξουμε από κοινού τους κανόνες. Είμαι βέβαιο και η χώρα μου και η κυβέρνησή μου είναι βέβαιη και πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει πρωτοπόρο ρόλο. Αλλά θα έπρεπε να είναι διεθνή η πρωτοβουλία από τον ΟΣΑ, το Παγκόσμιο Φόρουμ. Ε, είναι δανεική ε, φορεί για μια τέτοια πρωτοβουλία. Το Λουξεμβούργο όμω, επαναλαμβάνω, ε, δεν έχει κάνει τίποτε παράνομο και ήταν πάντα υπέρ ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού. Να πω επίση ολοκληρώνοντα ότι το Λουξεμβούργο έχει ήδη κάνει ε, την κατοίκον εργασία του ε, δίνοντας ε, τη λίστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άλλες αυτές τις αποφάσεις. Έχουμε και το σχετικό νομοθέτημα, έχουμε μια κεντρική επιτροπή για αυτά τα rulings από τον Ιανουάριο του 2015. Ετήσια δημοσιεύονται όλες αυτές οι αποφάσεις, άρα όλα είναι νόμιμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ριχσάρ Γιούγκ, τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πάμε προς την καλή κατεύθυνση, τουλάχιστον όσον αφορά την διαφάνεια. Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανταλλαγή στοιχείων και νομίζω ότι ακολουθούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η πρόταση του Πρόεδρου Ομπάμα να ζητήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις αμερικανικές, να μεταφέρουν τα κέρδη τους στις Ηνωμένε Πολιτείες και να φορολογηθούν εκεί με υψηλό συντελεστή είναι κάτι που νομίζω ότι ε, μπορεί να μας ικανοποιήσει. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει πρόεδρος όσον αφορά την εναρμόνιση της ε, φορολογίας. Και αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά υπονομεύει την ε, νομισματική μας ένωση δεν έχει νόημα να έχουμε κοινέ ε, πολιτικές όσον αφορά τα δημοσιονομικά, να έχουμε κοινό νόμισμα, ενώ η φορολογία κυμαίνεται από 10 έως 30% και όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές όσον αφορά τους συντελεστές, όσον αφορά τη βάση φορολόγησης και είπατε πολύ σωστά εσείς που εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι τα βήματα είναι πολύ αργά. Πρέπει λοιπόν, είναι δική μας ευθύνη, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόοδος. Όσον αφορά τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αυτό δεν είναι βέβαια κοινοτική αρμοδιότητα, είναι κάτι όμως που το πρότεινε η Γαλλία. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Και αν κάποιος ε, φαντάζεται μία τέτοια προσπάθεια να υπάρξει η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με πολύ χαμηλό συντελεστή και φανταστεί ότι για κάποια προϊόντα, κάποια παράγωγα παραδείγματο χάρη υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων opt-out γιατί κάποιες χώρες δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν αυτά τα προϊόντα καταλαβαίνετε ότι για τέσσερα χρόνια παραδείγματο χάρη μπορεί να υπάρξει η εξαίρεση, το opt-out και στο τέλος της τετραετίας να υπάρξει πραγματική εναρμόνιση για τις συναλλαγές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι και αλλιώς εδώ αναφερόμαστε στην συνεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε και τα τεκτενόμενα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Πορτογαλία. Ο Παύλο Άρα έχει το λόγο. Ε, eu pedi a Το δεύτερο τμήμα της συνάντησης. Ο κύριος Στόλογιαν έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ε, τα ίδια προβλήματα. Θα πρέπει να πληρώνονται οι φόροι και θα πρέπει να πληρώνονται εκεί όπου διεξάγεται ε, πραγματικά η οικονομική δραστηριότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειές της. Χαίρομαι γιατί το Συμβούλιο πράγματι κατέληξε σε μια κάποια συμφωνία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για τις σχέσεις ανάμεσα στην βασική τη μητρική εταιρεία και τις περιφερειακές εταιρείες για να μην υπάρχουν ε, καταχρήσεις. Τα κράτη-μέλη μπορούν να φορολογήσουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, στα εδάφη τους φυσικά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο όμως εσωτερικό. Υπάρχουν και άλλα εμπόδια, τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν μπορούμε να ορίσουμε σωστά εδώ και χρόνια. Σαν παράδειγμα, το μητρό των ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο μητρό, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ανώνυμες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, σε τρίτες χώρες, σε χώρες μέλη χωρίς να γνωρίζουμε τον πραγματικό του ιδιοκτήτη. Αυτό είναι ανυπόφορο. Φυσικά θα κληθούμε να συζητήσουμε και για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές συνήθως, οι οποίες αρνούνται να ενημερώσουν για τον τρόπο με τον οποίο πληρώνουν τους φόρους τους στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτω από τις συνθήκες αυτές να ορίσει κανείς σωστά και τη βάση επιβολής του φόρου. Θα πρέπει λοιπόν σε στενή συνεργασία και με τις Ηνωμένε Πολιτείες να καθορίσουμε ε, επίσης και τι ρυθμίσεις επιπλέον απαιτούνται για τους φορολογικούς παραδείσους και θα πρέπει οι χώρες αυτές να δεχτούν και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε διοικητικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει ε, να γίνονται συναλλαγές εμπορικές μη φορολογήσιμες. Σας ευχαριστώ. το Βελγικό Κοινοβούλιο, ο Ζορς ναι. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό που συζητούμε σήμερα. Είναι πολύ θετικό το ότι βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις συνειδητοποιούν πόσο επίγον είναι το θέμα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, με το ΦΑΤΚΑ η κυβέρνηση των ΗΠΑ πήρε πολύ σκληρά μέτρα και βεβαίως είδαμε ότι το θέμα της φόρο αποφυγής στην Ευρώπη από πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζεται σαν ένα δευτερεύον θέμα. Πρόκειται για κάτι το οποίο ουσιαστικά στερεί από κάποια ευρωπαϊκά κράτη από πολύ σημαντικές πηγές εσόδων. Βλέπουμε όμως ότι γίνεται ε, κατά κάποιο τρόπο ένας αγώνας για το ποιος θα είναι ο λιγότερο ε, αυστηρό στη φορολογία. Βλέπουμε ότι η Διερευνητική Επιτροπή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προχωρεί με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να το ξεπεράσουμε. Δεν στοχεύουμε μια συγκεκριμένη χώρα εδώ. Θέλουμε διαφάνεια. Χρειάζεται αυτοματοποιημένη ε, ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν ε, την φορολογία. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα φορολογείται εκεί όπου λαμβάνει η χώρα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι δίνουν πληροφορίες για αθέμητες ή παράνομες δραστηριότητες που αφορούν τη φορολογία. Και την ίδια ώρα θα πρέπει οι πρακτικές αυτές οι οποίες είναι αντιδεοντολογικές οι οποίες οδηγούν σε αυτόν τον επιθετικό φορολογικό ε, σχεδιασμό να καταδικάζονται. Πρόκειται για πρακτικές οι οποίες ναι μεν είναι πολλές φορές νόμιμες αλλά υπονομεύουν ε, την κρατική χρηματοδότηση. Και ξέρω ότι το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Εγώ γνωρίζω ότι γίνεται στο Βέλγιο. όπου οι πολυεθνικές μπορούν να ξεφύγουν από την ε, πραγματική φορολόγηση και εποφελούνται από εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νουέ από το, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα και τον ΩΣΑ και θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό παρόλο που υπάρχει το πρόβλημα και το εμπόδιο της ομοφωνίας για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις πρακτικές που επιτρέπουν σε κάποιες μεγάλες πολυεθνικές και ομίλους να μην ε, καταβάλουν τον φόρο που θα έπρεπε να καταβάλουν. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των ε, συμφωνιών ε, της φορολογίας, των tax ruling. Θα χρειαστεί χρόνος για να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Εν τω μεταξύ όμως θα μπορούσαμε ίσως να συμφωνήσουμε ότι κάποιες διατάξεις που δεν ε, βοηθούν την συνεργασία, όπως είπε και ο Βέλγος συνάδελφος, και που ουσιαστικά οδηγούν σε έναν φορολογικό ανταγωνισμό που αντιτίθεται στο πνεύμα ενός υγιούς φορολογικού ανταγωνισμού, όπως παραδείγμα χάρη κάποια υβριδικά σχήματα επιχειρήσεων που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις ευρωπαϊκές να έχουν ε, συνεδριάσεις του Διοικητικού τους Συμβουλίου στις Βερμούδες με μηδενικό συντελεστή φορολόγηση στη χώρα αυτή. Πρόκειται για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που τελικά καταφέρνουν να διαφύγουν και να μην καταβάλουν φόρο σε καμία απολύτως ευρωπαϊκή χώρα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κάλα Μετσκάλεφ από την Εστονία. Ναι, γεια σας. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα να δώσω αντίθετα εγώ θετικά παραδείγματα. Το 95% των, φορολο... των φόρων καταγράφονται ηλεκτρονικά και αυτό νομίζω ότι βοηθά ε, και καλό θα ήταν και άλλα κράτη να υιοθετήσουν την ηλεκτρονική φορολογική δήλωση. Τον Ιούνιο του 2014 θεσπίσαμε ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των τιμολογίων πάνω από 1.000 ευρώ για να καταπολεμήσουμε την φόρο αποφυγή και φοροδιαφυγή στο σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Από το Δεκέμβριο 2014 έχουμε τη νέα διαδικασία υποβολή φορολογικών δηλώσεων και με τον εταιρικό νόμο τον καινούριο είχαμε πολύ μεγαλύτερα ορθολογικά έσοδα της τάξης 47% μάλιστα με τον νέο ε, εταιρικό νόμο όπως είπα το Δεκέμβριο του 2014. Επίσης πέρυσι τον Ιούνιο υιοθετήσαμε επίσης και την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση με το Φρολικό Συμβούλιο για να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία και καταγράφονται πολύ πλέον, πάνω από 2% άτομα που δεν είχαν καταχωρηθεί πριν, τώρα είναι καταχωρημένα, είναι γεγραμμένα, έχουν φορολογικό μητρό. και μπορεί τα φορολογικά έσοδα να φαίνονται των 10 εκατομμυρίων ε, λίγα για κάποια άλλη χώρα και στην Ιστονία έχουν σημασία. Ο στόχος με όλα αυτά τα μέτρα ήταν να πετύχουμε κάποιους στόχους και αυτό και σας αναφέρω το θετικό και όχι αρνητικά που θα μπορούσαν να είναι κάποια παράπονα ή προβλήματα που έχουμε να επισημάνουμε. Ευχαριστώ. Ε, Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συνάδελφος Χάνα Μαλέτη της έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων όπως επίσης και τους Ευρωβουλευτές. Όλοι μας πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που τα ζητήματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, αλλά και ένα από τα βασικά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται σίγουρα για έναν τομέα που απαιτεί ενότητα, μια εναρμονισμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να έχουμε την οικονομική διακυβέρνηση, να έχουμε δομές συνεργασίας για το συντονισμό των δραστηριοτήτων. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλές ε, συνέργειες. Θα πρέπει να γίνουν επίσης επενδύσεις και στην εκπαίδευση των εφοριακών. Καλό θα ήταν να θεσπιστούν και νέα μέτρα για την ε, υιοθέτηση σωστών συστημάτων φορολογικής εποπτείας και παρακολούθησης. Θέλουμε σύγχρονες φορολογικές διοικήσεις που θα εντοπίζουν τα προβλήματα και θα τα αντιμετωπίζουν με επιτυχία. Πολλές φορές εφαρμόζονται εξατομικευμένα κάποιες προσεγγίσεις και αυτό είναι και πιο δαπανηρό. Αν είχαμε ένα ενοποιημένο σύστημα, θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσεις. Και θα έχει αυτό και ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους. Θα ξανακερδίζαμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας με αυτόν τον τρόπο. Και θα μπορούσε να δοθεί και όθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ από την Ιρλανδία. Πούμε. Ευχαριστώ. Κάποια από τα σχόλια που ήθελα να κάνω ακούστηκαν ήδη σχετικά με την φοροαποφυγή. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι χώρες ε, και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει ο ΩΣΑ. Νομίζω ότι εμείς ε, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα θέματα της φοροαποφυγής σε επίπεδο όσα από την άλλη πλευρά όταν τα συζητάμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμειγνύουμε και το θέμα της φορολογικής εναρμόνισης. Το θέμα της ε, εφαρμογής ενός σωστού φορολογικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο διασφαλίζει την ομιμότητα του συστήματος, ταυτόχρονα καθιστά τη χώρα ελκυστική σε επενδύσεις. Ενώ όταν μιλάμε για φοροαποφυγή είναι ένα θέμα το οποίο ε, πρέπει να απασχολήσει συνολικά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό. Σας ευχαριστώ. Φούξ από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι ο κοινό φορολογικός χώρος δεν είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν χώρες οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς σε πολλές χώρες. Είναι όμως ένας τρόπος ο οποίος θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο διαφορετικών ποσοστών επιβολής, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρώνουν με δίκαιο τρόπο τους φόρους τους, θα πρέπει όμως ταυτόχρονα άδικες ε, ρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας σε ορισμένες χώρες όπως το Λουξεμβούργο να καταργηθούν πλέον. Σχετικά τώρα με το ΦΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιβληθεί το σύστημα αντιστροφής ε, της απόδειξης εδώ. Έτσι θα βελτιώσουμε μόνο την συλλογή των φόρων αυτών. Σας ευχαριστώ. Σαχραντήλ από το από την Βουλή της Τσεχίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια πιο γενική παρατήρηση από, το, από ό,τι συνάδελφοι οι οποίοι προηγήθηκαν. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ξεκινώντας το γεγονός ότι το θέμα της επιβολής των φόρων είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι αποφάσεις ε, για το ε, επίπεδο επιβολής θα πρέπει να λαμβάνονται φυσικά σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η καταπολέμηση των φορολογικών απατών και της φοροδιαφυγής. Η καταπολέμηση σαν παράδειγμα των φορολογικών παραδείσων και να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο εσθονός συνάδελφος. Το πέρασμα στην ψηφιακή περιγραφή και σε των φόρων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που θα μας επιτρέψει να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα. Οι φορολογικοί πόροι ε, διασφαλίζουν τη σωστή ανακατανομή του πλούτου. Είναι κάτι το οποίο δεν το συζητήσαμε πάρα πολύ τουλάχιστον μέχρι τώρα. Υπάρχει μια ψευδέστηση θα έλεγα διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη και με το φυσικό δικαίωμα αν θέλετε στον πλούτο και στην ευημερία το οποίο θα έπρεπε να επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια ψευδέστηση αυτό, είναι κάτι το επικίνδυνο και καιρό είναι να αρχίσουμε να τα συζητάμε σε γενικότερο επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τελευταία παρατήρηση. Να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο έχει προτείνει και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης ήδη με τον πρόεδρο Γιούνκερ. Οι στόχοι πράγματι είναι υπερβολικά φιλόδοξοι. Να πολλαπλασιαστούν επί ε, τα, οι διαθέσιμες πιστώσεις ε, για επενδύσεις. Αυτό απαιτεί ε, μια αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και μια σωστή συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Όταν μιλάμε για ιδιωτικό τομέα σημαίνει και φορολογικά μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στον τομέα αυτό να επενδύσει. Σας ευχαριστώ. Από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο Σάση. Ευχαριστώ πολύ. Α, έζησε το μικρόφωνο σας. ΟΚ, να Μάλιστα, τώρα έργα δουλεύει. Ε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα ότι οι χώρες, μάλλον οι εταιρείε ε, θα πρέπει να πληρώνουν το ΦΠΑ εκεί που έχουν την οικονομική τους δραστηριότητα και να πληρώνουν μόνο μία φορά φόρους, όχι δύο φορές. Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός σήμερα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά για το μέλλον όχι, γιατί δεν θα έχουμε σε 10 χρόνια πια εταιρικό φόρο. Και γιατί θα συμβεί αυτό. Δείτε το τηλέφωνό μου. Το 5 με 10% είναι κόστος ε, κατασκευής. Όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδιασμός, μάρκετινγκ, προγραμματισμός. Αν ρωτήσετε πού γίνονται όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει. Γιατί μπορεί να γίνεται οπουδήποτε. Άρα είναι προς το συμφέρον μας, για παράδειγμα, σε αφορά τον προγραμματισμό ή το marketing, που είναι το μεγαλύτερο μέρος ε, της αλυσίδας. Να δούμε τι γίνεται, γιατί με την κατασκευή ξέρουμε ότι παραδείγματος γίνεται στην Ασία, ε, στις περισσότερες περιπτώσεις. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν. Έχουμε το πρόβλημα του φορολογικού ανταγωνισμού και τη φόρου αποφυγή. Υπάρχει ε, το λεγόμενο patent box στην Ολλανδία. Δηλαδή προσπαθούν όλε τι ευρεσιτεχνίε ε, να τι φέρουν στην Ολλανδία ε, και έχουν πολύ, πολύ, πολύ χαμηλού φορολογικού συντελεστέ. Τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον τώρα. Μπορεί πράγματι σε 10 χρόνια να μην έχουμε εταιρικό φόρο, άρα να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε Όμω, ε, να στήσουν ψηφίες θα πληρώνουν ένα 5% που δεν είναι πρόβλημα για αυτές και στο μέλλον όταν παρέχουμε υπηρεσίες επιχειρήσεις να πρέπει να πληρώσουν για αυτές τις υπηρεσίες οι εταιρείες και έτσι να, να χρηματοδοτηθεί η κοινωνία ουσιαστικά. Αλλά επαναλαμβάνω στο μέλλον δεν θα υπάρχει εταιρικό χώρος. Thank you. Last ο κύριος Λάγκεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Βεβαίως θα υπάρξει βάση του άρθρου 198 μια επιτροπή που θα κάνει τις απαραίτητες διαρευνήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι εδώ να συνδυαστεί η διερεύνηση αυτή με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και πραγματικά θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και αυτό σε πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, αυτό που συμβαίνει ε, στην ε, Ιρλανδία με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία, στις κάτω με το πώς αντιμετωπίζονται παραδείγματο χάρη κάποια ε, ιδρύματα. Κοιτάξτε πώς αντιμετωπίζουν, με τι ενιαίο τρόπο αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Βλέπουμε σήμερα ότι παρόλο που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ε, αποφάσεις ευρωπαϊκές, πριν από 15 χρόνια πήραμε αποφάσεις παραδείγματο χάρη για το θέμα του ΦΠΑ. Το Λουξεμβούργο συνεχίζει όμως και αντιμετωπίζει αυτές τις αποφάσεις σαν να μην υπάρχουν. Η φορολόγηση, παραδείγματο χάρη, είναι από 0,4 0,5. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένη παραβίαση της ε, αρχής του θεμητού ανταγωνισμού. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν. Ε, υπάρχουν συστάσεις, υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες αγνοούνται και βλέπουμε εδώ ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν μπει στην συναπόφαση αλλά και αυτά που έχουν μπει από τη συνθήκη του Άμστερνταμ στην, συναπόφαση συνεχίζουν να τα αγνοούν αυτά τα κράτη. Κοιτάξτε, η ψευδέστηση ότι ένα μικρό κράτος μπορούμε να το πιέσουμε και με αυτή την πίεση να πετύχουμε αυτά που θέλουμε, θα πρέπει να σταματήσει. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη τι γίνεται με την Ισπανία. Οι 25 μεγαλύτερες ισπανικές ε, επιχειρήσεις έχουν βάλει την έδρα τους που στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία. Μα σας παρακαλώ, ε, ας κοιτάξουμε τι γίνεται. Χρειάζεται φορολογικός ε, ανταγωνισμός, αλλά αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και επιβλαβής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το πρώτο τμήμα της ε, συζήτησης μας έχει ολοκληρωθεί. Συγγνώμη, δεν είδα ότι ζητήσατε το λόγο. Έχουμε κι άλλο ένα θέμα. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα και στον επόμενο κατάλογο μιλητών. Ζητώ συγγνώμη, δεν σας είδα. Και μπορώ να σας πω ότι αυτά που είπε ο κύριος Λάγκεν είναι λόγια πολύ ενδιαφέροντα. Τα γεγονότα είναι σαφέστατα. Άλλο είναι η εναρμόνιση και άλλο η φορολογική φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη. Και μεταξύ αυτών των δύο πρέπει να κινηθούμε, να λάβουμε μέτρα, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, και η διερεύνησή μας, η νομοθετική μας ε, πρωτοβουλία, η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι καθοριστική. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την συζήτηση για το θέμα αυτό, η οποία φυσικά δεν ολοκληρώθηκε και ε, καθ' τη διάρκεια του έτους θα συναντηθούμε πολλές φορές και ελπίζω να είμαστε σε θέση να πούμε ότι έγινε πρόεδρος. Περνάω στο δεύτερο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, που είναι το θέμα η ε, εποπτεία των ε, αρμόδιων αρχών στον τραπεζικό τομέα και το υπόλογο αυτών των αρχών. Έχει ξεκινήσει όπως ξέρετε η εποπτεία από μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με πολύ συγκεκριμένες και αυτές συνέπειες στον τομέα πώς ε, λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός πώς γίνεται ο απολογισμός ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συζητήσουμε τις προθέσεις μας, πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις αρμοδιότητές μας και πώς θέλουμε να υπάρξει και να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χούμπνερ. Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική πλευρά. Θα ασχοληθώ περισσότερο με θέματα νομικού τύπου. Αλλά δεν αρνούμε ότι η πολιτική διάσταση γενικότερα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης της ε, ε, Τραπεζικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όλα αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά θέματα. Ο δημοκρατικός έλεγχος είναι η καρδιά, αν θέλετε, της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια δημόσια ευρωπαϊκή πολιτική θεωρείται θεμητή εφόσον είναι έκφραση της λαϊκής βούλησης είναι μια προκαταρκτική αν θέλετε μορφή νομιμοποίησης της πολιτικής δράσης των ευρωπαϊκών οργάνων. Εφόσον βέβαια έχουν σαν στόχο να καλύψουν τις προσδοκίες και τους στόχους που θέτουν οι πολίτες. Αυτό ισχύει γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να δειχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την λεγόμενη εκ των προτέρων νομιμοποίηση υπήρξε ένα συμπλήρωμα στη συνθήκη το οποίο επικυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Οι αρχές της τράπεζας διορίζονται από τα κράτη-μέλη και επικυρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μιλάω. Και έχει επίσης και την εκ των υστέρων νομιμοποίηση, γιατί στην ουσία δημιουργεί το λεγόμενο δημόσιο αγαθό, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα σταθερό νόμισμα. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες δυσκολίες στα πλαίσια της καταμέτρησης του τρόπου και του ποσοστού ικανοποίησης το οποίο δίδει στους Ευρωπαίους πολίτες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό ακριβώς εμείς εδώ ελέγχουμε σε μόνιμη βάση την τράπεζα αυτή και η εμπειρία μας μέχρι τώρα δείχνει ότι ο έλεγχος αυτός σε επίπεδο πρακτικής είναι λειτουργικός. Αυτά για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα για τα θέματα της εποπτείας. Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας που ξεκίνησε από την προηγούμενο φθινόπορο έχει προσθέσει αν θέλετε ένα επίπεδο περιπλοκότητας στο θέμα του ελέγχου και του υπολόγου των εποπτικών αρχών. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε κάποιους δισταγμούς σε σχέση με τη νομική βάση της Τραπεζικής Ένωσης γιατί εξαίρεσε ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία συνομοθεσίας. Ένα άλλο θέμα ήταν ο διαχωρισμός της νομισματικής πολιτικής από τη μία και της εποπτικής δραστηριότητας από την άλλη. Οι εποπτικές αποφάσεις δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν τις αποφάσεις στο νομισματικό τομέα και τούμπαλι. Όλα αυτά συνδέονται και σε σχέση με τους διαφορετικούς στόχους του υπολόγου και του δημοκρατικού ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπόλογη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι εποπτικές αρχές είναι υπόλογες και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτό στην εισαγωγική του ομιλία. Τίθεται επίσης και το θέμα, αν θέλετε, των άνισων συνθήκων που επικρατούν στις χώρες ε, μέλη του ευρώ και στις χώρες μέλη εκτός ευρώ που θέλουν να συνεργάζονται σωστά με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχει συνεισφέρει θετικά για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν έχουμε λύσει συνολικά το θέμα βέβαια ε, και των φορολογικών θεμάτων που ασχολούνται, ε, που καλύπτουμε. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται πάντως από τις αρχές εποπτείας και από το σύστημα εποπτείας γενικότερα έχουν συνέπειες δημοσιονομικές. Και το δίλημα εδώ ήταν να υπάρξει ένας μηχανισμός εθνικού ελέγχου για το SSM χωρίς να δημιουργηθεί ένας επιπλέον κίνδυνος διασποράς και διάσπασης της εποπτικής διαδικασίας. Γι' αυτό λοιπόν οι ε, διαδικασίες οι εθνικές τώρα πλέον ε, εξελίσσονται σε εθνικό όπως είπαμε επίπεδο, δεν χρειάζεται να δώσω περισσότερες εξηγήσει. Υπό την αιγίδα λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας τίθεται πλέον ένα θέμα μιας νέας πρόκλησης αν θέλετε, καινοτόμου πρόκλησης μετά από την διαθεσμική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη μία και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την άλλη. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και για τον μηχανισμό εξυγίανσης. Γενικά υπάρχουν αρκετά χαίνοντα θέματα, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε στο να ελέγξουμε πλήρως το, πρόγραμμα, το πρόβλημα του ελέγχου και του υπολόγου των εποπτικών αρχών. Όλα θα εξαρτηθούν από την διαφάνεια με την οποία οι εποπτικοί μηχανισμοί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες τους. Μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Ναι, έτσι πιστεύω. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς ε, εξακολουθούμε να είμαστε αδύνατοι, θα έλεγα, σε σχέση, ανίσχυροι σε σχέση με τη νομική βάση. Ε, και αυτό το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με αλλαγή στις συνθήκες. Αυτή η αδυναμία δείχνει ότι απαιτήθηκε μια διακυβερνητική συμφωνία και για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα δουλειά η οποία πρέπει να γίνει εξαντλώντας τις πιθανότητες και δυνατότητες που δίδει η συνθήκη. Φερέιρα. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα λόγια που χρησιμοποίησε ο πρόεδρός μας Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση ήταν συνολικά μια επανάσταση είναι πολύ σωστά. Πράγματι δημιουργούμε κάτι εντελώς καινοφανές, κάτι που ήταν απαραίτητο και για πολλούς λόγους που τους γνωρίζουμε πολύ εξημών. Όμως βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία δημιουργίας της Ένωσης. Δεν είναι ολοκληρωμένη ακόμη. Όπως σας θυμίζω έχει τρεις πυλώνες η Τραπεζική Ένωση. Έχουμε ήδη ε, τους δύο ε, πρώτους, ε, την εννέα εποπτεία, την εννέα εκαθάριση, χωρίς να έχουμε το νέο σύστημα εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων. Και μέσα στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, όπως είπε και η Ντανούτα, ακόμη προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός προστασίας, backstop και να εφαρμοστούν στην πράξη διακυβερνητικές ρυθμίσεις. Στόχος μας τώρα είναι να καταλάβουμε η νομοθεσία και το νέο σύστημα σε ποιο βαθμό εξισορροπούν την ανάγκη να εγγυηθούμε αφενός την ανεξαρτησία του νέου οπτικού Συμβουλίου και του νέου Συμβουλίου Εκαθάρισης αφετέρου με την ανάγκη ύπαρξης ε, υποχρέωσης λογοδοσίας για να είναι νόμιμες οι αρχές αυτές. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω τι προηγήθηκε το Κοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερα δραστήριο για την οικοδόμηση της Τραπεζικής Ένωσης. Ήδη από το 2010 είχαμε ζητήσει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είχαμε επίσης ε, δραστηριοποιηθεί για τη δημιουργία των νέων εποπτικών αρχών, για να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των 28 μεμονωμένων εποπτικών αρχών που κάλυπταν τις συναλλαγές, ε, και τις πράξεις ε, των ε, μεσητών και των τραπεζικών. Δημιουργήθηκε οι τρεις αυτές αρχές για τη μοτοπιστική εποπτεία και θα μπορούσε να υπάρξει αντίρρηση, ένσταση για, την, για τον ορισμό των διοικητικών, των των συμβούλων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτές τις υποπτικές αρχές και επίσης ε, αυτές οι ευρωπαϊκές υποπτικές αρχές ήταν υπεύθυνες και έπρεπε να λαγοδοτήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από το 2012 μέχρι πρόσφατα εμβαθύναμε ακόμη περισσότερο στην κοινή κατανόηση, στην κοινή εποπτεία κοινή εκαθάριση εντός Τραπεζικής Ένωσης. Βασιζόμενοι σε αυτές, ε, στο παράδειγμα αυτών των ε, εποπτικών αρχών, αλλά προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο σε ένα κοινό επίπεδο. Οι αρμοδιότητες και δυνατότητες των εθνικών αρχών να περάσουν σε ένα ευρωπαϊκό φορέα. Και αυτό το καταφέραμε με μια σειρά μηχανισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει με ψυχοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και έπειτα στην Ολομέλεια τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στην επιλογή συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια πρώτη δηλαδή φάση άτυπων ακροάσεων και υπάρχει μια ακρόαση των υποψηφίων και η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα στην ΕΚΟΝ και μετά στην Ολομέλεια. Ο πρόεδρος επίσης του ενόπτου μηχανισμού πρέπει να έρθει στο Κοινοβούλιο να παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις και συμμετέχει και σε δημόσια ακρόαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του οπτικού μηχανισμού δις ετησίως. Μπορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει να γίνουν εμπιστευτικέ ακροάσεις για ειδικά θέματα που να αφορούν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων. Προφορικά επίσης αλλά και εγγράφος μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήματα προς τον ε, ε, αποπτικό μηχανισμό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συγκεκριμένα ο μηχανισμός αυτός παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ιστορικό των αποφάσεων που βέβαια είναι επιστευτικές αλλά είναι αποφάσεις που για μας είναι σημαντικές για να καταλάβουμε πώς έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος η διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Τώρα όλες αυτές τις διατάξεις τις έχουμε στον κανονισμό για τον νέο παπτικό μηχανισμό και όπως είπα υπάρχει και διοργανική συμφωνία που επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες αυτές. Τώρα προβλέπουμε ένα παράλληλο παρόμοιο σύστημα για τον νέο μηχανισμό εκαθάρισης. Είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της διοργανικής συμφωνίας που θα είναι λίγο πολύ κάτι αντίστοιχο με τον μηχανισμό τον εποπτικό. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σημαντικές βελτιώσεις ό,τι αφορά και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Ιδίω ό,τι αφορά την υποβολή ετήσια έκθεση από τα δύο συμβούλια. Αυτέ οι ετήσιες εκθέσει θα διαβιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχουσών κρατών μελών, ε, χώρων μελών τα κοινοβούλια αυτών των χωρών μελών μπορούν να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους και να τις υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα, τεχνικά κοινοβούλια πάντα, προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να διοργανώσουν ακροάσεις με τον πρόεδρο ή μέλος του Συμβουλίου του ε, Νεοποπτικού Μηχανισμού. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυξάνει τις εξουσίες και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ό,τι αφορά τη δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα αφού ε, είμαστε στη φάση της οργάνωσης του συστήματος ακόμα και βέβαια πρέπει να το εφαρμόζουμε και στην πράξη εν συνεχεία. Νομίζω και από αυτό ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε αυτή την υποχρέωση λογοδοσίας μεταξύ Ευρωπαϊκών, Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων, ώστε οι πολίτες να καταλάβουν ότι δεν μιλάμε για μια απόλυτη, απολυταρχική εξουσία. Σίγουρα είναι μια ανεξάρτητη εξουσία που όμως πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες και ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των πορτών που είναι οι εθνικοί και ε, οι, οι ευρωπαίοι βουλευτές. Θα σταματήσω εδώ. Αναλαμβάνω ότι είναι ένα τελείως καινούριο σύστημα, αυτό που δημιουργούμε τώρα. Και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συνειδητοποιήσουν ότι η ευθύνη πηγαίνει μαζί ακριβώς με αυτή τη νέα εξουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από το Κοινοβούλιο της Λετωνίας, ο Έντουαρτ Σμίθα. Ή, θα μιλήσω εγώ στη θέση του συναδέλφου, ο οποίος πήρε το λόγο στην αρχή της συνεδρίασης για το άλλο θέμα. Καταρχήν να σας πω ότι πραγματικά χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία αυτής της εποπτικής αρχής και όλους τους ε, κανόνες για να υπάρξει πραγματική διαφάνεια και λογοδοσία. Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητη αυτή η εποπτική αρχή και είναι πολύ σημαντικό κάποιος να έχει αξιοπιστία και θα πρέπει να στηρίξουμε αυτήν την φήμη και την αξιοπιστία αυτής της αρχής. Συμφωνώ με την κυρία Περέρα όταν λέει ότι πραγματικά η Τραπεζική Ένωση είναι ένα επαναστατικό βήμα καθότι ενισχύει την αξιοπιστία, τη φερεγγιότητα του τραπεζικού συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε αυτήν την ε, αξιοπιστία καθότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι τα κονδύλια αυτά βρίσκονται σε καλά χέρια. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να είναι ξεκάθαρο το ποιος είναι υπεύθυνο γιατί σε περίπτωση δυσκαλίας. Το θέμα της διακυβέρνησης, το θέμα της ανάκτησης. Ε, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πληγεί η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Ξέρετε ότι μια σημαντική τραπεζική κρίση χωρίς μηχανισμό προστασίας των πολιτών είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Το 2008 και 2011 δύο μεγάλες τράπεζες στην ε, Λετωνία κατέρευσαν, αλλά τότε ήμασταν σε θέση με ηρεμία να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας ε, για τους πολίτες μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο μηχανισμός με εναρμονισμένο τρόπο να εφαρμοστεί παντού σε όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Οι τρεις πυλώνες τώρα, ναι, μόλις τώρα ξεκινούν να λειτουργούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το εγχείρημα, το θέμα της εποπτείας είναι κάτι που μας απασχολεί ε, στα κοινοβουλιά μας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει από τη μία ο ανεξάρτητος χαρακτήρας αυτής της αρχής, από την άλλη να υπάρχει δυνατότητα λογοδοσίας και υποχρέωση λογοδοσίας και θα πρέπει αυτά τα δύο να είναι πολύ ισορροπημένα. Ευχαριστώ πολύ από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσατα ότι για να λύσουμε τα προβλήματα της κρίσης απαιτούνται κάποια έκτακτα και επίγοντα μέτρα και έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Μέτρα τα οποία θα χαρακτήριζα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας αυτό το ιστορικό αν θέλετε, αν θέλετε να επιμείνουμε στο θέμα ε, του ελέγχου και του υπολόγου των, ε, της Κεντρικής Τράπεζας και των ε, νέων θεσμών εποπτείας. Είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα το οποίο δημιουργήσαμε και αυτό δημιουργεί θέματα, αν θέλετε, ελέγχου. Να κάνω λοιπόν τώρα τρία μικρά σχόλια σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Πρώτον, έχει σημασία να διευκρινίσουμε ότι η έννοια της ανεξαρτησίας ενός πιστοτικού οργάνου ή και μιας κεντρικής τράπεζας και του ελέγχου του οργάνου αυτού είναι διακριτά μεταξύ τους αλλά και στενά συνδεδεμένα. Όσο πιο ανεξάρτητος είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός τόσο περισσότερο υπόλογος θα πρέπει να είναι. Υπάρχει δηλαδή ένας θετικός συσχετισμός ανάμεσα στα δύο αυτά χαρακτηριστικά και πρέπει να πούμε ότι μόνο εν μέρη έχει καλυφθεί η ανάγκη αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με άλλα λόγια, το επίπεδο ανεξαρτησίας είναι υψηλότερο από το επίπεδο ελέγχου. Δεύτερον, έχει σημασία να ξεκινήσει κανείς από ένα ειδικό χαρακτηριστικό της ε, οικονομικής αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η διαχειριστική τράπεζα σε επίπεδο εποπτείας, αλλά δεν έχει αναλάβει πλήρως τις εποπτικές αρμοδιότητες των χρηματοπιστωτικών αγορών σαν παράδειγμα, όπως το θέμα των κινητών αξιών, η διάρκεια, ε, η προστασία των καταναλωτών, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πάντα εθνικές αρμοδιότητες. Αυτή λοιπόν η μορφή ελέγχου του κινδύνου από τις τράπεζες που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται μια πλήρη εικόνα της λειτουργίας των μεμονωμένων τραπεζών. Απαιτείται μεταφορά πληροφοριών γι' αυτό και ακριβώς εδώ έγκυται και το επίπεδο δυσκολίας, γιατί υπάρχει δυσκολία στη σωστή ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών. Λοιπόν, βασικός μας στόχος τα επόμενα χρόνια είναι να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης όχι μόνο διαμεθοριακό αλλά και διατομεακό σε επίπεδο πληροφορίας. Είναι ένας βασικός στόχος εφόσον πράγματι θέλουμε να έχουμε ε, μια ισχυρή εποπτική διαδικασία. Τέλος, εφόσον πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, την ανάγκη δημιουργίας ενός προτύπου πρέπει να γίνονται σεβαστές τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, σωστός καθορισμός των κανόνων και των ευθυνών. Δεύτερον, πλήρης δημοκρατικών έλεγχος από το Κοινοβούλιο. Και τέλος, ισχυρότατη εντολή για εξωτερικούς ελέγχους, έτσι ώστε ε, να εγκρίνονται οι λογαριασμοί των τραπεζών αυτών και να εφαρμόζονται οι συστάσεις τους. Συνεπώς, αν γίνουν αυτά, θα έχουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό επίπεδο διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά απαιτούνται και άλλα ε, για να φτάσουμε στο επίπεδο ε, ελέγχου το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το θέμα δεν είναι μόνο να λαμβάνουμε στα πλαίσια αυτού του νομισματικού διαλόγου πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την εκπλήρωση της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το ποσοστό εκπλήρωσης αυτό. Πώς δηλαδή πετυχαίνει τους στόχους της η τράπεζα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της εντολής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και τις χώρες μέλη και το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν η ανεξαρτησία από τη μία και ο έλεγχος από την άλλη πρέπει να διασυνδεθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Καμπρίτα της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία που έχει τελέσει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ και την ε, κυρία Φερέρα. Και βεβαίω η πρόοδο που έχει επιτευχθεί είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την εποπτεία αλλά και την εκαθάριση. Βεβαίω θα πρέπει εδώ να ακολουθήσουν και οι εγγύησει των καταθέσεων. Ο τρίτο πυλώνας, τον οποίο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση ούτε να ξεχάσουμε ούτε να αγνοήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο τρίτο πυλώνας αν θέλουμε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Όταν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να μην ε, πληρώσουν τελικά οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ένα, μια παράλογη συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ξέρουμε σήμερα ότι οι πολύ σημαντικές ε, ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ε, καταρρεύσει, έχουν πτωχεύσει και εξαφανιστεί. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουμε εδώ την ε, λαϊκή δυνατότητα επιτήρησης, επέμβασης και φυσικά οι μεγάλες ε, ευρωπαϊκές τράπεζες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους ούτε να αναγκαστούν να έχουν μια συμπεριφορά και εδώ βεβαίως η αρμοδιότητα είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα εποπτείας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίσει τους μηχανισμούς δημοκρατικού ελέγχου. Ξέρετε ότι και μία πορτογαλική τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία εκαθάρισης. Σήμερα μια επιτροπή συνοδεύει αυτήν την διαδικασία. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος λοιπόν είναι καθοριστικός και αυτό ισχύει και σε εθνικό επίπεδο αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως να δραστηριοποιούμαστε τα πλαίσια όλων των ε, οικονομικών οργάνων, κοινοβουλευτικών επιτροπών, με συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, έτσι ώστε αυτός ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας να απολογηθεί για το πώς έχει η κατάσταση και είναι πολύ διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εργασία σας. Ναι, θα προσπαθήσουμε να μην ξεχνάσουμε αυτόν τον τρίτο πυλώνα που πολύ σωστά εντοπίσατε. Ο κύριος Νεοφίτου από την Κύπρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χρηματοπιστωτική κρίση μας έδωσε την ευκαιρία στην Ευρώπη να διορθώσουμε λάθη αρχιτεκτονική στην Ευρωζώνη. Η Τραπεζική Ένωση έπρεπε να είχε από καιρό γίνει, όπως και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Εν πάση όμως περιπτώσει ε, εμείς λέμε στα, ελληνικά κάλλιον αργά παραποτέ. Όμως δεν είναι αρκετό το ότι δημιουργήθηκε η Τραπεζική Ένωση, το ότι έχουμε πλέον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Το κυριότερο είναι να βρούμε τους μηχανισμούς οι τράπεζες να είναι τράπεζες. Να μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη και την οικονομία μιας χώρας. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει πως οι τράπεζες δεν εξασκούν αυτό τον ρόλο. Γι' αυτό και δύσκολα θα φύγουμε από την ύφεση να πάμε στην ανάπτυξη. Και γίνεται μια δημόσια συζήτηση κατά πόσον θα αυξήσουμε και πάλι τα δημοσιονομικά ελλείμματα για να πετύχουμε την ανάπτυξη που είναι ένας λάθος δρόμος την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να τη στηρίξουν οι τράπεζες χρηματοδοτούντες βιώσιμες ε, επενδύσεις. Θέλω να κλείσω κύριε Πρόεδρε με ένα προβληματισμό. Ε, προέρχομαι από την Κύπρο όπου έχει επευληθεί για πρώτη φορά στην ιστορία την οικονομική της παγκόσμιας κοινότητας και όχι μόνο της ευρωπαϊκής το κούρεμα καταθέσεων. Και μένει ένα ερώτημα στο να απαντήσουμε ε, χωρίς ακόμα να έχω καταλήξει προσωπικά το ποιο είναι το πιο δίκαιο και το πιο σωστό ε, τα λάθη των τραπεζών να τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι φορτώνοντας επιπρόσθετο δημόσιο χρέος για τα λάθη των τραπεζών ή είναι πιο δίκαιο τα λάθη των τραπεζών να τα πληρώνουν κατά κύριο λόγο οι μέτοχοι, οι καταθέτες και οι κάτοχοι αξιογράφων. Είναι μια συζήτηση που θα διαρκεί για πάντα χωρίς να υπάρχει η τέλεια απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Πάλο Σα. Από την ε, συνελευτή Πορτογαλίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Αστικών Κοινοβουλίων, η απάντηση στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 οδήγησε στο να καταβάλουν υψηλότατο τίμημα οι λαοί πολλών χωρών και για να σώσουν την αξιοπιστία τους τα κράτη-μέλη προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν την ψευδέστηση ότι με τις νέες ε, διατάξεις για εποπτεία ε, δικαιολογούνται, δικαιολογούνται οι αφεμάξεις από το δημόσιο και τομέα. Δεν λύνονται όμως τα προβλήματα με παραπάνω εποπτεία. Το δείχνει η κατάσταση στην Πορτογαλία για έξι χρόνια. Εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιήθηκε για τη διάσωση μιας τράπεζας. Οι εποπτικοί μηχανισμοί υιοθετήθηκαν με νομοθέτημα. Το 2014 όμως το πρωτογαλλικό κράτος χρειάστηκε να δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 4 δι συγκεκριμένα δημόσιο κονδυλίων για να σώσει τις τράπεζες για μια ακόμη φορά. Δεν χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση των ε, ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Απλά θα πρέπει οι αποφάσεις της Ένωσης να μην βασίζονται στα συμφέροντα των ε, πολύ μεγάλων τραπεζών και των πολυεθνικών, γιατί αυτό θα είχε άκρο αρνητικέ επιπτώσει που θα οδηγήσει και στην απώλεια εθνική κυριαρχία ε, στην νομισματική και δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη θα αναγκαστούν να, συνεχίσουν σε αυτό τον φιλελεύθερο δρόμο. Η Πορτογαλία όμως πρέπει να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία στον τραπεζικό τομέα που είναι στρατηγική σημασία για την οικονομία μας. Πρέπει να είμαστε ε, στην υπηρεσία και ε, των συμφερόντων του καλού του πορτογαλικού λαού. Ο Έχουμε αυτό το μηχανισμό, τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει σωστά αλλά και δημοκρατικά. Ο Ντέιβις από τη Βουλή των Λόρδων έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα κάνω ερώτηση και δεν γνωρίζω την απάντηση. Έχω την εντύπωση όμως θα πρέπει να εστιάσουμε στην ερώτηση αυτή. Τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις και η δράση της ε, ελληνικής κυβέρνησης έχουν δημιουργήσει έλλειψη εμπιστοσύνης, έχουν υπονεωμεύσει την εμπιστοσύνη όλων προς ε, την ε, ελληνική κυβέρνηση, τη δράση της, το χρέος και τη στάση όσον αφορά αυτούς που κατέχουν ε, την ελληνική, το ελληνικό χρέος. Το πρόβλημα λοιπόν του κόστους του κεφαλαίου, των επιτοκίων, η φόβη ότι θα συνεχιστεί αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης και ότι θα αυξηθεί μάλιστα, κινδυνεύει η κρίση να ξεπεράσει την Ευρώπη, να ξεπεράσει την Ελλάδα και να υπάρξει, όπως ξέρετε, περαιτέρω διαφυγή κεφαλαίων εκτός Ευρώπης. Εάν υπάρξει πτώχευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε μία ακόμα πιο τρομακτική κατάσταση. Κάποιος θα πρέπει εδώ να είναι υπεύθυνο ε, υπεύθυνο ε, σε αυτή την περίπτωση είναι καταρχήν το εθνικό κράτος, κατόπιν η Ευρώπη και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία τελικά δανείζει και παρεμβαίνει. Είναι δυνατόν όμως σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αντικαταστήσει όλα αυτά τα κονδύλια, όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία έχουν διαφύγει έτσι ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ζώνη του ευρώ, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή ενδεχομένως θα αποφασίσει να πτωχεύσει το ελληνικό κράτος. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί μια απόφαση η οποία στο πιο δραματικό σενάριο θα είναι να κλείσουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, να απαγορευθούν όλες οι κινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επαναλαμβάνω, είναι αυτή που δανείζει σε, τελική, σε τελικό βαθμό. Δεν είναι αυτή που θα πρέπει αρχικά να παρεμβαίνει για να λύνει αυτά τα προβλήματα. Τι θα γίνει λοιπόν σε μια τέτοια τραγική κατάσταση, σε ένα εφιαλτικό σενάριο, αν αυτό συμβεί και μπορεί να συμβεί κατά την άποψή μου. Βλέπουμε εδώ τους πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί εμείς οι πολιτικοί είμαστε αυτοί που τελικά πρέπει να προστατεύσουμε το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. και Κινέ ναι, από το Βέλγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν απέχει τόσο μακριά ήδη και ακόμα μάλλον στοιχίζει πολύ για τα δημοσιοοικονομικά και έχουμε την εντύπωση ότι ορισμένοι θεωρούν ότι ολοκληρώθηκαν οι μεταρρυθμίσεις. Τροποποίησεις έγιναν πράγματι. Πάνω στο να δούμε ποιο ασκεί έλεγχο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όμως οι βασικές μεταρρυθμίσεις που είχαν προβλεφθεί ιδίω στο τέλος της προηγούμενης ε, νομοθετικής περίοδου, η λεγόμενη μεταρρύθμιση μπαρνίε είναι κάτι για το οποίο δεν γίνεται πλέον λόγος, ε, πιστεύω πια. Δηλαδή, τι συμβαίνει με την απαγόρευση χρηματοπιστωτικών πρακτικών που είναι πολύ ρυψοκίνδυνες ε, και γίνονται από ορισμένες τράπεζες. Τι γίνεται με το διαχωρισμό των τραπεζικών καθηκόντων τι γίνεται με το συστημικό κίνδυνο των τραπεζικών ιδρυμάτων για την οικονομία των κρατών μελών. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το πρωί μιλήσαμε για τις επενδύσεις Juncker. Αλλά και τα τραπεζικά δρήματα, οι καταθέσεις, οι αποταμίσεις έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν σε όλα αυτά. Φαίνεται όμως σήμερα να μην έχουν όλα αυτά σημασία για τους εθνικούς δομοθέτες ούτε για τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη και θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα αυτό σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, έχει εγκαταληφθεί εντελώ η φιλοδοξία να έχουμε ακόμα βαθύτερε μεταρρυθμίσει σε σχέση με αυτέ που έγιναν από τότε που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική τραπεζική κρίση. Θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά πλέον σήμερα. Νομίζουμε ότι είναι όλα ρόδινα ξανά. Και αν πιστεύουμε έτσι, εγώ νομίζω ότι αναλαμβάνουμε τεράστιο ρίσκο. Πράγματι, η απόφαση της ΕΚΤΑ για τη λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, μπορεί να βοηθήσει τις χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία και πάλι όμως. Πρέπει όλα αυτά να περάσουν ε, υποχρεωτικά τις τράπεζες. Είναι αυτή η καλύτερη λύση? έχουμε πολλά ερωτηματικά. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο αίτημα δεν θέλει κάποιο άλλο να δώσει το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ελίζα Φερέιρα. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ πλούσια η συζήτηση. Ήταν πραγματικά πολύ πλούσια η συζήτηση. Δύο νομίζω τα ζητήματα που, κατα... που έγιναν σαφή. Το πρώτο είναι ότι έχουμε ένα νέο σύστημα πια, το οποίο αναπτύσσεται, εξελίσσεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα του Λόρδου Ντέιβις. Όπως είναι το τρέχον πλαίσιο, η ΕΚΤ υποτίθεται ότι δεν μπορεί να καλύψει τραπεζικές απώλειες, όμως είναι γεγονό ότι όταν θα ισχύει πλήρως τραπεζική ένωση και θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά την 1η Ιανουαρίου πλήρως και ε, ο μηχανισμός εκαθάρισης, μιλάω για το Γενάρη του επόμενου έτους, δεν έχουμε ολοκληρώσει με το σύστημα εκαθάρισης. έχουμε τον εποπτικό μηχανισμό προς το παρόν. Τότε όμως από το 16 και μετά η απόλυση των τραπεζών ε, θα είναι κάτι που θα επομίζονται οι ιδιοκτήτες της τράπεζας κάθε. Και θα πρέπει να συνεχίσει υπό διαφορετικό καθεστώς το καλό κομμάτι της τράπεζας αυτό είναι καθάριση και όχι κήρυξη μια τράπεζα αφαιρέγγια. Ως αφαιρέγγιας. Θα υπάρχει λοιπόν ένα ταμείο, θα το χρηματοδοτούν οι ίδιες οι τράπεζες με βάση το προφίλ τους και άρα η τράπεζα θα πληρώνει. Δηλαδή θέλουμε να συγκρατήσουμε τις απώλειες εντός τραπεζικού τομέα και να μην τις μετακυλήσουμε στην ΕΚΤ ή στο φορολογούμενο σε τελική ανάλυση. Όμως, ε, σε μια άλλη κατάσταση, εκροή καταθέσεων κάτω από 100.000 ε, ευρώ, το είπε και ο Κύπριος βουλευτής. Πράγματι λοιπόν, εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα νέο εποπτικό σύστημα με τους ίδιους κανονισμούς, με μια εποπτεία που δεν γίνεται σε εθνικό αλλά σε υψηλότερο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό δηλαδή επίπεδο. Και αν έχουμε και δυνατότητα εκαθάρισης ταυτόχρονα, ο καταθέτης ουσιαστικά θεωρεί, θα πρέπει να θεωρεί ότι τα κεφάλαιά του είναι εγγυημένα και στην τράπεζα αλλά και στην τράπεζα Β, εφόσον διέπονται και οι δύο από τους ίδιους κανόνες, την ίδια εποπτεία, τους ίδιους ε, μηχανισμούς εκαθάρισης. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν αυτή τη σταθεροποίηση της κατάστασης και πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα τα οποία, οποία αναφερθήκατε πολλοί συνάδελφοι. Ένα άλλο στοιχείο, απατώντας τον Παουλ Σα και περνάω στα πορτογαλικά. Είπατε Ποιες ελευθερίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Άρα χρειάζεται ένα κοινό σύστημα κανόνων για τη ρυθμίση των τραπεζών και την εποπτεία των τραπεζών. Αλλά χρειάζονται και κοινοί κανονισμοί και μηχανισμοί εκαθάρισης, ώστε οι μέτοχοι της τράπεζας να απομίζονται το κόστος και το βάρος του ρίσκου που αναλαμβάνουν. Πρέπει να αλλάξει η τραπεζική κουλτούρα ουσιαστικά και όχι φορολογούμενοι να είναι αυτοί που διασώζουν τις τράπεζες μέτοχοι. Θα πρέπει λοιπόν οι τράπεζες να έχουν ένα ταμείο, να έχουν κονδύλιο προς αυτό. Και νομίζω ότι έτσι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερη σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα. Ο Πάολο επίσης πολύ σωστά τα είπε Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανεξαρτησίας και λογοδοσίας. Με ένα κοινό σύστημα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι τράπεζες ε, στην Ευρώπη θα έχουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως του σε ποιο κράτος μέλος έχουν την έδρα τους. Να μην έχουμε επίσης μια υπερβολική συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος στο κέντρο των χωρών. Γι' αυτό όμως θα απαιτηθούν περαιτέρω εξελίξεις. Θα πρέπει οι ε, εποπτικές αρχές και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχουν έντονη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Το 2010 εμείς στο Κοινοβούλιο ζητήσαμε να υπάρξει μια κοινή κουλτούρα, μια κοινή νοοτροπία, θέσπιση κοινών κανόνων στην εσωτερική αγορά των 28 κρατών. Τώρα λοιπόν, με περικοπές πεπολογισμών στις αρχές αυτές ή με άλλα ε, μέσα, το θέμα είναι να μην έχουμε αφενός το τραπεζικό, της Τραπεζική Ένωση που θα είναι πάρα πολύ επιτυχημένο το σύστημα και εκτός να υπάρχει πλήρης αστάθεια και αποσταθεροποίηση η ενίσχυση λοιπόν και του εξωτερικού αλλά και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το δίκτυο ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφοριών. Είναι βασικός στόχος για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Καμπρίτο για το σχόλιο το οποίο έκανε. Θεωρώ, Εντοάρντο, ότι το σύστημα ως έχει μπορεί να λειτουργήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρήζει ενίσχυσης. Αυξάνεται το επίπεδο εποπτείας και αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε μεν θετικό, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στους επόπτες και στους εποπτευόμενους έτσι ώστε να υπάρχει και σωστή ενημέρωση αυτών οι οποίοι εποπτεύουν, αναλαμβάνουν τη διαδικασία της εποπτείας. Για τον Γάλλο συνάδελφο, ο οποίος αναφέρθηκε για τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε σχέση ε, με τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το έχουμε υπόψη μας αυτό, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας Έχουμε ένα εισηγητή και δύο σκιώδεις. Η διαδικασία όπως σας είπα συνεχίζεται. Η έκθεση έχει πλέον, η πρόταση έκθεσης έχει ολοκληρωθεί. Η συζήτηση των τροπολογιών θα, δίνει την, θα γίνει την 23η Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στις 24 Μαρτίου. Επαναλαμβάνω, η διαδικασία συνεχίζεται. Τα θέματα αυτά έχουν σημασία για το Κοινοβούλιο. Σας ζητώ να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν είναι ίσως τόσο δημοφιλές, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση ε, δείχνει ότι πρέπει να υπολογίζουμε πολλά, γιατί οι αλλαγές οι οποίες έγιναν σε επίπεδο θεσμικών αλλαγών έλυσαν ορισμένες δυσκολίες, διατηρούνται όμως ορισμένες ε, ε, δυσκολίες στην περίπτωση κατά την οποία μια πολύ μεγάλη Ευρωπαϊκή Τράπεζα αντιμετωπίσει προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται ε, και στις Ηνωμένε Πολιτείε με τον λεγόμενο κανόνα Βόλκερ και στη Μεγάλη Βρετανία με τον κανόνα Ρίκερ και γενικά να ωφεληθούμε από τις εμπειρίες των υπολείπων χωρών. Δεν θα πρέπει να απορρίψουμε αυτά τα οποία έχουμε πετύχει, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες ε, σε επίπεδο λεπτομέρειας διαφοροποίησεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να κλείσει η συνεδρίασή μας. Νομίζω ότι έγιναν δύο πλούσιες συζητήσεις, δύο τμήματα και οι δύο συζητήσεις έδειξαν την ανάγκη η οποία χρειάζεται για σωστή συνεργασία. Ιδιαίτερα το δεύτερο θέμα, το θέμα της ε, εποπτείας και του ελέγχου των εποπτικών αρχών, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις γύρω από το SSM δίνουν την δυνατότητα ελέγχου στις χώρες μέλη αλλά πρέπει να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών έτσι ώστε να, καταστήσουμε τον ενιαίο μηχανισμό ακόμα πιο ελέγξιμο και ε, υπόλογο. Συνεπώς λοιπόν η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί πλήρως την ταχύτητα των αλλαγών και δεν συνειδητοποιεί πλήρως επίσης την ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού και αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού. Πρέπει να είναι ισχυρός ο μηχανισμός αυτός, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, αλλά πρέπει να λειτουργεί πάντα στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου. Και έτσι θα αυξήσει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη της τραπεζικής βιομηχανικής δραστηριότητας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 2.45 στην Ολομέλειά μας. Ευχαριστώ.